Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν με μεγάλες προσδοκίες. Περιμένουν πάρα πολλά πράγματα από την Ευρώπη και περιμένουν ένα ισχυρό μήνυμα από μας αύριο. Θερμά χειροκροτήματα. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη που προβλέπει την έκθεση του κυρίου Κάρες για τη Συμφωνία της Βασιλείας 2 και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Θα ξεκινήσω δίνοντα το λόγο στον κύριο Κάρας για τέσσερα λεπτά, που είναι και ο συγγετής. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Κύριε Καράς, έχετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχει στόχο την ε, διαμόρφωση θέσης για τις διαπραγματεύσεις ε, της Επιτροπής της ε, Βασιλείας και έχουμε βεβαίως κάποιες απαιτήσεις προς την ε, Κομισιόν για το σχέδιο οδηγίες. Παρά το ότι και εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συγητές, παρά το ότι λοιπόν στην Επιτροπή εγκρίθηκε η έκθεση με 38 έναντι 0 αρνητικών ψήφων, ένιωσα την ανάγκη να καταθέσω και εγώ κάποιες τροπολογίες ως ηγητής. Τρεις αναφέρονται στις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα εντωμεταξύ στην Βασιλεία και άλλες τρεις ε, στις, ε, στις προδιαγραφές ρευστότητας. Θεωρούμε πως δεν είναι σωστό να περάσουμε αυτομάτως ε, από το 2018 στον πρώτο πυλώνα το leverage ratio, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία αξιολόγησης. Δεύτερον, στις προδιαγραφές ρευστότητας υπάρχουν κάποια ανοιχτά ε, σημεία τα οποία πρέπει να συζητηθούν για να είμαστε απολύτως επίκυροι. Κυρίε και κύριοι, απορώ λίγο για τα κράτη, για τα κράτη μέλη της Ένωσης στην Βασιλεία τα οποία αξιολόγησαν την διαδικασία ως ολοκληρωμένη, παρά το ότι κατά την άποψή μας δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και ε, αμερικανικών τραπεζικών δομών, ούτε ίση όροι ανταγωνισμού μεταξύ της κλασικής τραπεζικής λιανικής και των επενδυτικών τραπεζών και ταυτόχρονα δεν έχουμε ορισμό ορισμό της ρευστότητα. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως η κρίση κατέδειξε πως ε, χρειαζόμαστε μια αλλαγή του πλαισίου και λογικό είναι βεβαίως να το δούμε αυτό το ζήτημα και να υποβάλουμε προτάσεις. Αλλά η κρίση επίσης κατέδειξε πως πρώτα απ' όλα έχουμε μια κρίση ρευστότητας και όχι μια χρήση ιδίων κεφαλαίων. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα ίδια κεφάλαια. Στη Lehman Brothers, παραδείγματος χάρη, τα ίδια κεφάλαια ήταν 11% και κατά την άποψή μας είναι πέντε τα σημεία τα οποία είναι ανοιχτά. Πρώτον, δεν υπάρχει μελέτη επιπτώσεων για το τι θα σημαίνουν τα συμφωνημένα για την ανάπτυξη, για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ αυτό να το κάνει και να το υποβάλει άμεσα η Κομισιόν. Δεύτερον, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το σορευτικό αποτέλεσμα όλων αυτών των κανόνων που διαβουλευόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή Βασιλεία 3, προδιαγραφές ε, της ε, ρευστότητας, φόρος χρηματοπιστωτικέ συναλλαγές, έκτακτη εισφορά στι τράπεζε κτλ. Δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμοί π.χ. όσον αφορά την ερμηνεία αυτών των ε, διατάξεων και όσον αφορά βεβαίω το ποιο θα είναι το περιθώριο εισαγωγή. Κατόπιν δεν υπάρχει διαφορά δεν υπάρχει μάλλον ίδιας ορισμός του κεφαλαίου όσον αφορά τις τράπεζες Λιανικής και τις επενδυτική τράπεζες, καθώς επίσης και τον λόγο μόχλευσης μετά τι αποφάσει της Αμερικής. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν υποβάλει πρόταση οδηγίας η Κομισιόν και δεν πρέπει να ολοκληρωθούν μετά τους, ε, πριν τους G20 αλλά πριν από την Βασιλεία. Αλλιώς θα μείνουμε θεατές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρνιέ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ισηγητά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Λίγες μέρες μετά την ε, υπογραφή της συνθήκης της Βασιλείας και την αποδοχή της χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία εδώ να συζητούμε ενώπιον του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι είναι πρωταγωνιστή στην παγκόσμια σκηνή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ ε, τον κύριο Κάρας για όσα μας είπε και θα ήθελα ε, να τον ευχαριστήσω και για τα σημεία κριτικής τα οποία ανέφερα και τα οποία βεβαίως εντελεχώς θα συζητηθούν και θα μελετηθούν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμμερίζομαι κύριε Κάρας την ε, ε, άποψή σας σχετικά με την υπογράμμιση ε, των ειδικών στοιχείων της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας. Η ανάγκη αξιολόγησης επιπτώσεων και μάλιστα σε βάθος και βεβαίως όλα τα θέματα που άπτονται του ανταγωνισμού και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η καλύτερη κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών είναι απαραίτητη έτσι ώστε το χρηματοστατικό σύστημα να γίνει πιο σταθερό και πιο ισχυρό αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει κυρίες και κύριοι βουλευτές και το γνωρίζετε άλλωστε γιατί ε, δουλεύετε πάνω σε αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη επιτήρηση, καλύτερη και αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση, ε, προστασία απέναντι στην κερδοσκοπία, δυνατότητα αντιμετώπισης και πρόληψης βεβαίως των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών κρίσεων. Πολλά έχουν γίνει ε, μέχρι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως ε, και με τη βοήθειά σας ε, το νέο σύστημα υποπτίας, η πράσινη βίβλωση για τη διακυβέρνηση και βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική της πλευρά κάνει τη δικιά της δουλειά και με τρόπον ώστε μέχρι τα τέλη του, της επόμενης άνοιξης να έχουμε υποβάλει και σε εσά και στο Συμβούλιο το σύνολο των κειμένων που είναι απαραίτητες έτσι ώστε ε, να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση στη διάσκεψη κορυφής των 20. Ε, και βεβαίως προτάσεις και σχετικά με την ε, επιβλέψη και σχετικά με το short selling. Θα ήθελα σήμερα να ασχοληθώ ε, με τα τρία θέματα τα οποία απασχολούν και τον ε, κύριο Κάρας. Ε, πρώτα απ' όλα τις εγγύησεις όσον αφορά τις τράπεζες, τις συνεταιριστικές τράπεζες όσον αφορά το Time Warren Capital αυτό ε, θα μας δώσει την ε, δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας τις δυνατότητες αυτών των μη εισηγμένων ε, τραπεζών οι οποίες όμως λειτουργούν στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Αυτή τη στιγμή συζητούν και μελετούν τα θέματα αυτά ε, οι εμπειρογνώμονες. Δεύτερον, όσον αφορά την ρευστότητα καθώς επίσης ε, και το λεγόμενο liquidity buffer, ρυθμιστικό αποθεματικό ρευστότητας για την Δανία και για την Αυστρία όντως έχουν εκφραστεί πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις από την Επιτροπή και γι' αυτό ακριβώς δεν έχει ακόμα εξευρεθεί συμφωνία επί του θέματος αυτού. Έχουμε επιφυλάξεις και οι υπηρεσίες μας σε συνεργασία με τους εταίρους μας της Βασιλείας θα ε, συνεχίσουν ε, να ε, ασχολούνται με το θέμα των covered bonds. Τρίτον, ε, όσον αφορά τις ε, ε, δεσμεύσεις των G20 πρέπει να πούμε ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τις συμφωνίες της Βασιλείας, κυρίως δε όσον αφορά το θέμα της περίοδου παρακολούθησης του πυλώνα 2 εν ώψη της παγωγής σε μεταχείριση πυλώνα 1. Αυτό το ανέφερε και ο κύριος Κάρας και είναι εξαιρετικά θετικό στοιχείο. Δύο λόγια να πω τώρα σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας της Βασιλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλά μαθήματα θα πρέπει να μάθουμε από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση η οποία ταρακούνησε όλο τον κόσμο και η οποία κατέδειξε ότι δεν ήταν αρκετά οπλισμένη η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Ε, η νέα Συμφωνία της Βασιλείας προστίθεται στην ε, προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει κινήσει όσον αφορά την ενίσχυση του οπλοστασίου μας ε, για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους, ε, ε, τέτοιου είδους προβλήματα. Τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει μέχρι τώρα οδεύουν προς την κατεύθυνση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και σε αυτήν βεβαίως συμβάλλει η νέα συμφωνία της Βασιλείας. Είναι φυσικό επακόλουθο το γεγονός ότι βεβαίως θα δοθεί, μια, θα δοθεί η δυνατότητα βαθμίας εξηγή ε, του ε, τραπεζικού συστήματος καθώς επίσης ε, και θα δοθεί και η δυνατότητα στι επιχειρήσει βαθμιαία να προσαρμοστούν έτσι ώστε να μην αποσταθεροποιηθεί το οικονομικό σύστημα στα πλαίσια της βασιλείας θέλουμε να έρθουμε και σε συμφωνία με τις τρίτες χώρες και στην, στην επόμενη διάσκεψη της ε, Σεούλ την 20η Νοεμβρίου ε, θα ασχοληθούμε ε, σε επίπεδο G20 με το θέμα αυτό. Βεβαίως λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εθνικούς κανόνες αλλά φυσικά ε, οι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έστω και αν ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητά της. Ε, φυσικά θα κάνουμε και μικροοικονομικές και μακροοικονομικές αναλύσεις της Συμφωνίας της ε, Βασιλείας και για τα αποτελέσματα θα σας πληροφορήσουμε και εσάς κύριε Κάρας αλλά και τους συναδέλφους σας. Όσον αφορά την εφαρμογή θα αρχίσει να ισχύει από το πρώτο τρίμηνο του 2011 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2013. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να παραμένουμε ε, ε, ε, παραμένουμε λογικοί. Βεβαίω είναι καλό βήμα η συμφωνία της Βασιλείας, αλλά θα πρέπει μαζί με όλες τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προχωρήσουμε έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε τις σοβαρές βλάβες που άφησε πίσω της η χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, να προχωράμε με μικρά βήματα έτσι ώστε να κάνουμε την αυτήν την βασική μεταρρύθμιση με τρόπο σωστό και παρακολουθώντας αυτά που και οι εταίροι μας είτε οι Ηνωμένε Πολιτείε είτε άλλες χώρες εφαρμόζουν. Τέλος, συμφωνώ με τον ε, κύριο Κάρα. Συμφωνώ κύριε Κάρας μαζί σας ότι ε, θα πρέπει να ε, ε, ενισχυθεί η θέση και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία αυτή. Γι' αυτό ακριβώς δεσμεύομαι να αναφέρομαι ενώπιον της Ολομελίας σας για όλες τις μελλοντικέ εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εκ μέρου των πολιτικών ομάδων τώρα, πρώτα απ' όλα ο κύριος Γοζές έχει το λόγο εκ μέρου του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πολύ σύντομα. Θέλω πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το εξαίρετο έργο του συναδέλφου μας Κάρας. Ήμουνα κι εγώ από εκείνου που θέλησαν να έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλία πριν να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι αναγκαίε διατάξει για να εφαρμοστεί η Συμφωνία τη Βασιλεία. Η δουλειά που έκανε λοιπόν ο συνάδελφο Κάρα με τη συνεργασία βέβαια των σχεδόν εισηγητών μα ε, οδήγησε να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό που γνωρίζετε και που δεν θα επαναλάβω. Εννοείται ότι συμφωνώ με όσα είπατε και με την αποφασιστικότητά σας ώστε η ρύθμιση αυτή να είναι αποτελεσματική και ρεαλιστική και πάνω απ' όλα σε διεθνές επίπεδο να μην δημιουργήσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τώρα για να έρθω στο θέμα μας αυτό καθ' αυτό. Διαπιστώνω ότι συχνά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα λόγια που ακούμε επίσημα και στην πραγματικότητα που ακολουθεί. Διαπιστώνουν επίση ότι χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε για παράδειγμα, έχουν την κακή συνήθεια να κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο εμεί δουλεύουμε, ενώ εκείνοι οι ίδιοι δεν εφαρμόζουν τι διατάξει που θα έπρεπε να εφαρμόσουν. Πιο συγκεκριμένα για τη Βασιλεία, είναι ζωτική σημασία οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να τυχαίνουν ίση μεταχείριση και να μην υποβάλλονται σε κυρώσει από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε τις ε, τράπεζες που κανονικά υποβάλλονται στην Βασιλεία, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Σας υπενθυμίζω ότι εγκρίθηκε τον Ιούνιο για τη διακυβέρνηση των Αμερικανικών Δημοσιονομικών. Όμως στην πράξη δεν έχει προχωρήσει το πράγμα. Δεν τίθεται σε εφαρμογή διατάξεις τελικά που όμως εφαρμόζουν άλλες ε, οντότητες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω λοιπόν κύριε Επίτροπε να φροντίσετε να μην υπάρξει στρέβλωση ανταγωνισμού σε βάρος των γαλλικών τραπεζών, των ευρωπαϊκών τραπεζών και γενικότερα σε βάρο εκείνων που χρηματοδοτούν την οικονομία. Εννοείται ότι οι τράπεζε πρέπει να έχουν τον κύριο ρόλο που έχουν, που είναι να ενισχύσουν την οικονομία, αλλά δεν πρέπει από την άλλη μεριά να του επιβάλλουμε υπέρμετρε κυρώσει. Ευχαριστούμε κύριε Γκοζέσλη πρόεδρο. Ο κύριο Μπούλμαν τώρα, για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να διαπιστώσω κάτι. Η Επιτροπή της Βασιλείας είναι ένα φόρουμ ε, λίγο πολύ έξυπνων κεντρικών τραπεζιτών και εποπτικών αρχών αλλά δεν έχει και το αλάθητο και οπωσδήποτε δεν νομοθετεί. Ο νομοθέτης κύριε Επίτροπε βρίσκεται εδώ. Το ξέρετε και εμείς ξέρουμε ότι το ξέρετε. Και ο νομοθέτης αυτός θα φροντίσει να δει τι θα έρθει επιτάπητος και αν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Οπωσδήποτε θέμε οι διατάξεις κεφαλαιακών απαιτήσεων να ενταθούν. Βλέπετε που έχουμε φτάσει. 20-30% του ΑΕΠ έχει υποθηκευτεί για να σώσουμε τις τράπεζες. Οπωσδήποτε αναμένει ο κόσμος να λάβουμε τα μέτρα μας για να μην ξαναβρεθούμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Οπωσδήποτε θέμε και εμείς να υπάρχουν αντικυκλικά στοιχεία σε αυτή την διασφάλιση των τραπεζών όπως έχουν ληφθεί επί σειρά ετών στην Ισπανία και έπρεπε βεβαίως βλέπετε να έρθουμε σημερινή κατάσταση για να αποδειχθεί πόσο σωστά ήταν γιατί δεν έκαναν χειρότερο τραπεζικό σύστημα αλλά πιο εύρωστο όμως υπάρχουν βασικά ερωτήματα και ευχαριστώ τον κύριο Κάρας για το ότι τα βασικά αυτά ζητήματα είναι στο κέντρο της έκθεσής του, την οποία υποστηρίζουμε πλήρως. Πρώτα απ' όλα, ναι, πράγματι, χρειαζόμαστε μία μελέτη επιπτώσεων, η οποία θα είναι πολύπλοκη και θα μας λέει πρώτα απ' όλα ποια θα είναι η επίπτωση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά οπωσδήποτε και στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή τι θα γίνει από εδώ και μπρο με τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, την διαβεβαίωση πως αυτή τη φορά τα συμφωνηθέντα θα εφαρμοστούν και σε άλλες επικράτειες. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό πριν νομοθετήσουμε. Αλλιώς πάλι ασυμμέτρια θα, θα έχουμε, όπως στο παρελθόν. Και τρίτον, δεν μπορούμε να έχουμε διακριτική μεταχείριση νομοθετικών φορμών. Αυτοί οι οποίοι απέδειξαν το σωστό τους ρόλο κατά τη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή αυτοί οι οποίοι βοήθησαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες και δεν ασχολήθηκαν μόνο με διασυνοριακούς κινδύνους, δεν πρέπει να τιμωρηθούν και από πάνω επειδή ήταν πιο εύρωστοι. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν διασφαλίζεται. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση και να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε και πρακτικά κάτι τέτοιο. Γιατί οι τράπεζες έχουν μεγάλη αξία βεβαίως όταν λειτουργούν σωστά και πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον. εάν εφαρμόσουμε αυτά τα οποία από ό,τι φαίνεται προβλέπονται στη Βασιλεία που δεν επιτρέπεται να είναι η τελευταία λέξη που θα αποδεχτούμε. Πρέπει λοιπόν να μετρηθούν αυτά τα μέτρα ως προς το εξής. Να διασφαλίζουν την ίδια ποιότητα χωρίς διακρίσεις, να είναι ευέλικτα ως προς τον ε, τρόπο εκπλήρωσης και βεβαίως αηφόρα. Αυτή είναι η ε, αφετηρία από την οποία ξεκινάμε. Θέλουμε οπωσδήποτε να περιοριστεί η μόχλευση και να εκτιμηθεί το προφίλ κινδύνου όπως ε, το θέλει και η Κομισιόν και ελπίζουμε βεβαίω και στην συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Μπούλμαν. Τον λόγο έχει η κυρία Μπόουλς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Όταν ε, συζητήσαμε γι' αυτό και είπε ότι μοιάζει με την ελβετική γραβιέρα, γεμάτη τρύπε. Πράγματα δηλαδή πολλά θα ξεφύγουν. Οι τράπεζες συζητάνε για τη Βασιλεία 3. Όλοι έχουν ε, στο στόμα τον όρο εθνικές διατάξεις, εθνικές εξαιρέσεις κλπ. κλπ. Μόλις αποφασιστεί ένα πλαίσιο για την εναρμόνιση και την σταθερότητα, τότε αρχίζει η προσπάθεια να φτιαχτούν οι τρύπες, τα παραθυράκια. Έχω βαρεθεί. Γιατί αυτή η Ευρώπη πρέπει τελικά να είναι το χαμένο παιδί της Βασιλείας. Δεν θα έπρεπε. Δεν ήταν αυτή η αρχική πρόθεση της Βασιλείας Τρία. Και η G20 ήταν ξεκάθαρη. Οι τράπεζε θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίζουν κρίσεις σαν και αυτήν που μόλι είχαμε. Και το κεφάλαιο είναι σημαντικό να υπάρχει έτσι όπως πρέπει. Να μην τα βάζουμε με την πραγματική οικονομία. Όπως κι άλλοι, περιμένω μακροοικονομικές ε, αξιολογήσεις. Όχι μόνο για τη Βασιλεία, αλλά γενικότερα για δημοσιονομικούς κανονισμούς μετά τη Βασιλεία που εσεί και ο Επίτροπος ε, Ρεν μου υποσχεθήκατε όταν ήρθατε εδώ για τις ακρόασεις. Τελικά όμως δουλεύετε στα μυστικά και κρατάτε απόρριτο για τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς επεκτάθηκε η διορία για την Βασιλεία και αυτό φτάνει. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε να δεχτούμε. Τα μέτρα ρευστότητας, κύριε Επίτροπε, δεν έχουν λυθεί πλήρως. Και εγώ θέλω περισσότερα κίνητρα. Να μην υπάρχει αυτή η συγκέντρωση όπως υπάρχει τώρα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να σκεφτούμε και να μην επαναλάβουμε τα ίδια ε, μέτρα, οπότε και τα ίδια λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν και τώρα με τα εποπτικά μέτρα και να καταστρέψουμε έτσι και την πραγματική οικονομία μέσω επενδύσεων κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φιλίπ Λαμπέρτς τώρα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα η Βασιλεία 3 θα, ε, θα πρέπει να είναι βάση εργασία και όχι την μέγιστη περίμετρο ε, που μπορεί να ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτοί που λένε εάν προχωρήσετε ακόμα περισσότερο ε, την Βασιλεία τότε θα υποφέρει η ανταγωνιστικότητα των τραπεζών μας. Και εγώ απαντώ ότι αυτό που μας ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η βιωσιμότητα των ε, επιχειρήσεών μας. Ε, επίσης, τα κράτη-μέλη, όταν, ε, συγγνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν μπορούν και όποτε δουν ότι τα καταφέρνουν, προχωρούν μόνες τους. Εμείς λοιπόν γιατί δεν μπορούμε. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι τα 8 χρόνια τα οποία αναφέρονται εδώ είναι υπερβολικά και επίσης δεν έχει προβλεφθεί ότι όσον αφορά την κατανομή ε, των μερισμάτων και των μπόνους ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Είναι απαράδεκτο, ε, είναι, δεν είναι καθόλου σοβαρό οι τράπεζες από την μία πλευρά να λένε ότι έχουν προβλήματα οικονομικά ενώ από την άλλη πλευρά ανοίγουν τα ταμεία τους για να πάρουν μπόνους τα στελέχη τους επίσης για τις τράπεζες οι τράπεζες οι οποίες παραπονιούνται ότι δεν θα έχουν πλέον τις δυνατότητες και τα περιθώρια κέρδους που είχαν τα χρυσά χρόνια. πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί που δουλεύουν στη βιομηχανία αυτοί δηλαδή που δουλεύουν στην πραγματική οικονομία έχουν περιθώρια 2-3% και δεν τρέπονται γι' αυτό. Επομένω, θα πρέπει να καταλάβουν το πάρτι τελείωσε και ότι θα πρέπει και αυτοί να προσαρμοστούν σε αυτά τα ε, ε, ε, ποσοστά κέρδου. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ. Γνωρίζω πως δεν έχει τελειώσει η οικονομική κρίση και χρειαζόμαστε περαιτέρω δάνεια από τις τράπεζες. Βλέπουμε όμως στην Ιρλανδία την προηγούμενη εβδομάδα πως ακόμα ζητάνε διάσωση από το φορολογούμενο οι τράπεζες. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να αναλαμβάνουν κίνδυνο, αλλά χρειάζονται κεφάλαιο και ρευστότητα για να μπορούν να αντέξουν όταν υπάρχει πρόβλημα με αυτό το κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Βεβαίως η έκθεση του κύριου Κάρας είναι μέρος μόνο της λύσης. Είναι σαφές από τον αριθμό τροπολογιών πως οι ευρωβουλευτές θέλουν να δουν τις λεπτομέρειες και τον αντίκτυπο. Και πρέπει το ίδιο να γίνει και για τις εγγυήσει ε, στα παράγωγα. Η πρώτη λοιπόν ε, αξιολόγηση αντικτύπου έγινε στη Βασιλεία αλλά είναι εμπιστευτική. Οπότε οι τράπεζε πρέπει να την δώσουν στη δημοσιότητα και να τη χρησιμοποιήσουν. Και όταν κάνουμε διεθνείς συμφωνίες πρέπει να ισχύουν παγκοσμίω. Όχι μόνο εδώ και στη Wall Street, παγκοσμίω υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο. Η ρήτρα 24, η ρήτρα 40 που περιγράφει τα ομόλογα. Ναι, η 43 πρέπει να δει την στήριξη των ε, μικρών τραπεζών η Βασιλεία, αλλά όπως το βλέπω εγώ στα αγγλικά, είναι πως από ό,τι φαίνεται εμείς προκαταλαμβάνουμε το συμπέρασμα που θα βγάλουν. Επιπλέον ε, έχουμε συμφωνήσει πως θα μεταβούμε σε ένα δεσμευτικό λόγο μόχλευσης. Ας μην απομακρυνθούμε από αυτό. Συμφωνώ πως εκεί όπου υπάρχουν σωστές τοπικές πρακτικές πρέπει να συνεχίσουν, αλλά στις εξετάσουμε δημοσίως και όχι να φέρνουμε εξαιρέσεις από το παράθυρο γιατί η αγορά θα υποθέσει πως υπάρχει έτσι ένα παραθυράκι για να προωθήσουμε τις λανθασμένες και όχι σωστές πρακτικές. Ευχαριστούμε κύριε Θόρτου. Περνάμε τώρα στους άλλους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα κυρία Λούλινγκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας, τον κύριο Κάρας, για την εξαίρετη δουλειά του. Τον υποστηρίζω απόλυτα, την προσέγγιση του δηλαδή και την προβληματική του. Παρ' όλα αυτά θέλω να υπογραμμίσω στα δύο λεπτά που έχω στη διάθεσή μου ένα θέμα το οποίο θίγεται στην έκθεση και που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο. Έχει να κάνει με τις εγγυήσεις όσον αφορά τη ρευστότητα που έχουν οι τράπεζες. Το πρόβλημα με τη ρευστότητα στην Ευρώπη που θέλουμε να επανακαθορίσουμε εδώ θα έπρεπε να εξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, νομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες. Είναι κάτι που πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα και οι επενδύσεις που γίνονται ε, πρέπει να τις βλέπουμε ευρέως. Η σημερινή όμως πρόταση της Επιτροπής της Βασιλείας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και δυσανάλογες πάνω στην ευρωπαϊκή οικονομία, αν συγκρίνουμε με το τι γίνεται σε άλλες μεγάλες οικονομικές ζώνες στον κόσμο, όπως για παράδειγμα νομένες Πολιτείε. Εννοείται ότι χαιρετίζω την συμφωνία του Ιουλίου της Βασιλείας που αναγνωρίζει τις συγκητικές αυτές επιστολές σαν ενεργό κεφάλαιο για την κάλυψη ρευστότητας. Όμως, παρόλα αυτά, ζητάω και από την Επιτροπή της Βασιλείας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Μισελ Μπαρνιέ, στο οικονομικό αυτό μέσο, όργανο, να δώσετε μεγαλύτερη αναγνώριση ώστε να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη διαφοροποίηση όσον αφορά το ενεργητικό και να αποφύγεται στρεβλώσει στην αγορά. Είναι ένα οικονομικό μέσο που δεν ελοχεύει κινδύνους και άρα μπορεί να ευνοηθεί η εξέλιξή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λούλιν. Κύριε Ποδηματά τώρα το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή συζήτηση για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η Επιτροπή της Βασιλείας είναι ένα ακόμα βήμα το οποίο υπαγορεύτηκε από την πρόσφατη κρίση. Μια κρίση που κατέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο ελλείψεις και αδυναμίες στη ρύθμιση και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποδόμησε το κυρίαρχο τότε δόγμα της αυτορύθμισης των αγορών και ανέδειξε την ανάγκη η αυστηροποίηση των κανόνων τόσο για την κεφαλαιακή επάρκεια όσο και για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. μέσα σε αυτό το κλίμα η επιτροπή της βασιλείας κατέληξε σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει ορισμένες βασικές αρχές ορισμένες βασικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στους κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας για να θωρακιστεί καλύτερα το τραπεζικό σύστημα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής στην ευρώπη η έκθεση του συναδέλφου του κυρίου κάρας αναδεικνύει πολλές σημαντικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη όπως είναι η ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς όπου το 80% της διανοδότησης στηρίζεται στα πιστωτικά ιδρύματα η ανάγκη εκδημοκρατισμού της διαδικασίας της βασιλείας μεταξύ των άλλων και με την ενεργότερη συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και ε, βεβαίως η πρόταση για την συμπερίληψη του συνόλου των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης στα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης ώστε να περιορίζεται ο αντίκτυπος των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. θέλω ωστόσο να επαναλάβω ότι τα νέα μέτρα για την κεφαλαιακή υπάρκεια συνιστούν μια μίνιμουμ αναθεώρηση και εξακολουθούν να απαιτούνται μεταρρυθμίσεις γενικότερου χαρακτήρα με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. η ευρώπη το είπε ο κύριος επίτροπος έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με την υιοθέτηση του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας αλλάζουμε το τοπίο και προωθούμε τον ενισχυμένο συντονισμό ως ένα βασικό εργαλείο πρόληψης. δεν πρέπει ωστόσο να μείνουμε εκεί χρειάζεται να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα με τη θέσπιση εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου φορέων που ως σήμερα λειτουργούν ανεξέλεγκτα όπως είναι οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου ή οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων. χρειάζεται στη βάση των προτάσεων που παρουσιάσατε πρόσφατα κύριε επίτροπε να προχωρήσουμε σε κανόνες για τη ρύθμιση συναλλαγών που παρουσιάζουν σημαντική αδιαφάνεια και ως εκ τούτου αυξημένο συστημικό κίνδυνο όπως είναι η αγορά των εξωχρηματιστηριακών παραγόγων και των ακάλυπτων πωλήσεων. και τέλος κύριε επίτροπε επειδή αναφερθήκατε στη σεούλ στη σύνοδο του g 20 χρειάζεται να ηγηθούμε της προσπάθειας για τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όχι βεβαίως για να εκδικηθούμε ή για να τιμωρήσουμε τις τράπεζες αλλά για να περιορίσουμε την κερδοσκοπία και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες της ένωσης που σήμερα πληρώνουν το τίμημα της κρίσης ότι μεριμνούμε για να υπάρχει μια δικαιότερη κατανομή των βαρών. Euh, Ευχαριστούμε κυρία Ποδηματά. Ο κύριος Κλίντς τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αν πρέπει να κρατήσουν περισσότερο κεφάλαιο οι τράπεζες, τότε αυξάνεται και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε απώλειες. Δυστυχώς όμως η Βασιλεία, η Επιτροπή της Βασιλείας δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ε, τραπεζών που είναι σημαντικές για το σύστημα. Χαιρετίζω λοιπόν ε, την πρόταση του κυρίου Κάρας να ληφθεί υπόψη το μέγεθος και η παγκόσμια δικτύωση τραπεζών για να έχουν υψηλότερες απαιτήσεις αυτές οι τράπεζες. Διαφοροποιημένα επίσης πρέπει να δούμε την μόχλευση του χρέους. Ε, μόνο εάν διαπιστωθεί πως ε, δεν οδηγεί σε αρμπιτράζ και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού θα πρέπει να σκεφτούμε μία υποχρεωτική ρυθμίση αυτού του μέσου. Θα πρέπει όμως ό,τι κάνουμε να ισχύει παγκοσμίω. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επηρεάζουν οι Αμερικάνοι το ότι γίνεται στη Βασιλεία και μετά να μην τα εφαρμόζουν κιόλα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και θα δούμε εάν και κατά πόσο θα επιτύχουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίτρας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω πως είμαι ικανοποιημένος για το ότι το Κοινοβούλιο προετοίμασε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα λοιπόν τον εισηγητή την τελευταία δεκαετία είδαμε πρωτοφανείς εξελίξεις ε, νέων ε, χρηματοπιστωτικών μέσων ε, που έκριναν την φύση σήμερα των χρηματαγορών. Οπότε από πλευράς υποπτίας πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε αξιόπιστη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στις χρηματαγορές. Τώρα, τα μέσα αυτά έχουν γίνει τόσο πολύπλοκα ώστε είναι αδύνατον ε, για τις ε, εποπτικές αρχές να ελέγξουν αυτά τα μέσα. Πρέπει να θυμόμαστε και βεβαίως την παγκοσμιοποίηση των χρηματαγορών οπότε η εποπτεία η καθίσταται αναποτελεσματική. Η ανάπτυξη λοιπόν των ε, χρηματοπιστωτικών αυτών οργανισμών σημαίνει πως ε, και η εποπτεία καθίσταται πιο δύσκολη. Οπότε υπάρχει η έλλειψη μιας γενικής εικόνας ε, του τομέα. Οπότε, πρέπει να εστιάσουμε στην ασφάλεια του συστήματος και οι τωρινές ε, συμφωνίες της ε, Βασιλείας αφορούν την ε, κεφαλιακή επαρκιά και χαίρομαι για το ότι είδαμε τα ζητήματα της ρευστότητα και των αντικυκλικών κινήσεων. Όσον αφορά τώρα την αποτελεσματικότητα του λόγου του δίκτυ κεφαλαίου νομίζω πως η τυποποίηση αυτών των λόγων είναι κάτι το θετικό γιατί θα μας επιτρέψει να σώσουμε τις τράπεζες. Ευχαριστούμε ο κύριος Λέντινγκσον τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ θετικό το ότι η δουλειά για τους νέους ιδίως πόρους προχωράει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα για να πετύχουμε την οικονομική σταθερότητα. Η πρόταση έχει διατυπωθεί. Θέλω όμως να επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα, τα οποία θα ήθελα να είναι πιο ξεκάθαρα για μένα. Φυσικά και είναι σημαντικό να μην πιέζουμε πολύ τις τράπεζες. και να μην ε, βάλουμε ένα πολύ μικρό χρονικό πλαίσιο για την ε, συμμόρφωσή τους. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να πάμε και πολύ αργά. Ο στόχος μας πρέπει να είναι οι τράπεζες να έχουν αρκετή σταθερότητα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επόμενη οικονομική κρίση. Όμως, να μιλάμε για το 2017-2018 δεν ξέρω πόσες τράπεζες θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Χρειάζεται συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλες περιοχές του κόσμου. Η φιλοδοξία μας πρέπει να είναι ολόκληρος ο τραπεζικός τομέας να είναι σταθερός, όχι μόνο ένα κομμάτι του τραπεζικού αυτού τομέα. Εκεί όπου υπάρχει αδύναμη ρύθμιση ή όπου η ρύθμιση προχωράει αργά, θα μπορούσε να πλήξει και όλους τους υπόλοιπους. Έπειτα, οι δοκιμές αντοχής βοηθούν για να ξέρουμε κατά πόσο είναι σταθερή μια τράπεζα. Όχι, βοηθάει δηλαδή σαν μηχανισμό πέρα από τις κεφαλαϊκές απαιτήσει που έχουμε βάλει. Πρέπει να είναι κριτήριο. Το μέτρο πρέπει να είναι κάτι που να μπορούμε να μετρήσουμε και να μπορούμε και να βελτιώσουμε. Ο οικονομικός τομέας πρέπει να ξέρει ότι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σμίτ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, νομίζω ότι είναι καλύτερα, είναι όντως μια καλή εξέλιξη ε, αυτή η σχετική με την Βασιλεία. Όμως ε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ε, ότι τελικά δεν δυναμητίζουμε, μάλλον δεν κυρώνουμε περαιτέρω τις δραστηριότητες μικρού κόστους γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες συναλλαγές τουλάχιστον στο σκανδιναβικό τραπεζικό σύστημα σύστημα. Ε, επομένως λοιπόν ε, κάποιες ε, αποφάσεις της βασιλεία μπορεί να είναι καλές αλλά καμιά φορά η ισορρευτική αποτίμηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εάν οι νέοι αυτοί τραπεζικοί κανόνες αρχίσουν να εφαρμόζονται θα πρέπει να ξέρουμε τελικά έχοντας κάνει κάποιες μελέτες επιπτώσεων που θα μας οδηγήσουν γιατί καμιά φορά το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Τώρα, ο κύριος Καντσιάν έχει το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε. Κύριε Καντσάν. Αλλάξτε μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεστε καλά. Υπάρχει κάποιος, κάποια αντίχηση που γίνεται. Τώρα με ακούτε. Ωραία. Ναι, ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε ε, πολύ τον ε, συνάδελφο Κάρας γιατί έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Εμείς αδύναμοι παρακολουθούσαμε αυτήν την ε, σφαιρική παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση Μερικοί είπαν μάλιστα ότι θα μπορούσαν να είχαν τα πράγματα ακόμα χειρότερα από ό,τι τελικά πήγαν. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και εσείς κύριε Επίτροπε ε, οδηγείτε μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει στην σταθερότητα και στις απαραίτητες εγγύησεις λαμβάνοντας ε, υπόψη ότι ε, η οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει και στην ε, διάσωση της Ευρώπης είναι πολύ σωστό το ότι συζητούνται, συζητάται η απαγόρευση των ακάλυπτων πωλήσεων ο φόρος για τις τραπεζικές συναλλαγές και βεβαίως περιμένουμε την τελευταία λέξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως κύριε Επίτροπε να είστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην περάσουμε περάσουμε όπως συμβαίνει καμιά φορά από τη μία άκρη ε, στην άλλη από το ένα άκρο μάλλον στο άλλο ε, δηλαδή να μην οδηγηθούμε τελικά σε μέτρα τα οποία θα ανακόψουν ε, την οικονομική ανάπτυξη γιατί μην ξεχνούμε ότι παραμονεύουν πάντα οι δυσκολίες και η γραφειοκρατία και η νομική βραδύτητα χρειαζόμαστε ανάπτυξη ανάπτυξη και πάλι, και πάλι ανάπτυξη όπως έλεγε προημερών σε αυτήν την αίθουσα ο πρόεδρος Μπαρόζο. Βεβαίως ξεκινούμε μία οδό την οποία θα πρέπει να ε, ξεκινήσουμε όλοι με μεγάλη ε, αίσθηση ευθύνης ε, αλλά να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να προστατεύσουμε και το τραπεζικό σύστημα κυρίως δε να προστατεύσουμε τις μικρές τράπεζες, τις συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη εγκύτητα με τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε τώρα με το Catch the Eye. Ο πάλι πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ. Νομίζω πως όλοι συμφωνούν πως πρέπει να διασφαλίσουμε την εντοχή του τραπεζικού στήματος και χάρη στον κύριο Κάρας γνωρίζουμε πως δεν είναι ίση η του ανταγωνισμού οπότε δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε έτσι και υπάρχει ο κίνδυνος να βάλουμε αυτογκόλ Και πρέπει βεβαίως να τονίσουμε πως η ΕΠΑ και η Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικές. Ε, η ΕΠΑ βασίζονται στις χρηματαγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις των τραπεζών να δίνουν δάνεια. Και το βλέπουμε στην Ιρλανδία που δεν μπορούν πλέον να δανειοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, είναι μια χαρά βιώσιμες χρεοκοπούν γιατί έχουν στερέψει τα δάνεια. Οπότε διασώζουμε από τη μία τις τράπεζες ε, και χρηματοδοτούμε και τις, ε, τα μπόνους και τις ε, χρυσές συντάξεις και αποζημιώσεις των στελεχών τους. Οπότε με ενθαρρύνουν αυτά τα οποία είπε εδώ πέρα ο κύριος Επίτροπος πως θα προσπαθήσει να επιφέρει μια ισορροπία να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού και τότε επιτέλους αντί για αυτόν κολ θα βάλουμε και εμείς κανένα γκολάκι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη. Τον λόγο έχει ο Επιτροπός Μπαρνιέ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε και βεβαίως ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές που πήραν το λόγο. Τους ευχαριστώ για τις προτάσεις τους, ε, για την ενθάρρυνσή τους και για όλες τις παρατηρήσεις τις οποίες βεβαίως με προσοχή έχουν γράψει τα μέλη της ομάδος μου και ο κύριος Σμιτ και ο κύριος Κλίντς και ο κύριος Λουτφίνσον ε, και ο κύριος Κέλλης πριν από λίγο ε, το θέμα της στόχευσης, ε, της σωστής στόχευσης. Ναι, βεβαίως θα θέλουμε η στόχευση να είναι καλή και μάλιστα σε τρία σημεία. Πρώτον, η ζυγοστάθμιση κατά κάποιο τρόπο της ίδιας της συνθήκης της Βασιλείας γιατί βεβαίω, βάσει της συμφωνίας της Βασιλείας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η δεύτερη προσπάθεια ε, στάθμισης ε, είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας της διάσκεψης των 20 γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή ε, η στάθμιση και ο κύριος Κέλλης προηγουμένως είπε πολύ σωστά αναφέρθηκε στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, και ε, βεβαίω ξέρουμε ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τράπεζες χρηματοδοτούν το, τις επιχειρήσεις και την οικονομία πολύ περισσότερο από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε και το τρίτο, ε, και εδώ λέω στον κύριο Λαμπέρτς, ότι ναι, ε, και το κάνουμε πριν από τις Ευρωπαϊκές, ε, πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας βλέπω κύριε Λάμπερτ, δεν με παρακολουθούσατε. Λέω λοιπόν ότι χωρίς να περιμένουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνουμε μέτρα θα πηγαίνω στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και ε, ε, πηγαίνω και μιλάω με όλους τους υπευθύνου έτσι ώστε να μιλάμε για όλα τα θέματα. Για τη Βασιλεία 1, 2, 2,5, 3, 4 και επίσης και για άλλα πολύ ευαίσθητα θέματα τα οποία ενδεχομένως ε, μπορούν να αποτελέσουν και σημείο ε, ε, διαφοροποίησης με τις ΗΠΑ συγκεκριμένα τα λογιστικά συστήματα Ε, γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ε, ενώπιον σας ότι πραγματικά εμείς θα ε, κάνουμε αυτές τις τρεις σταθμίσεις και επαναστοχεύσεις. Έχετε δίκιο κύριε Καντσάν σε αυτό που λέτε ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και καμιά φορά τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να, αποβληθούν. να ε, ε, αποβούν μοιραία ε, για την ανάπτυξη και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Άκουσα επίσης τον βουλευτή ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μελετών. Μα κύριε Μπιλμαν βεβαίως έχετε δίκιο έτσι, έτσι πρέπει να κάνουμε και βεβαίως εμείς εδώ στο Συμβούλιο θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν το αφήσουμε στα χέρια της Βασιλείας. Βεβαίως εμείς ε, θα κάνουμε όλες αυτές τις μελέτες με το CRD4 έτσι ώστε πριν ξεκινήσει καν η συζήτηση να έχουμε συγκεκριμένες ε, συζητήσεις. Η ε, κυρία Μπόιλς, βεβαίως έχετε δίκιο όταν λέτε ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν είναι business as usual. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και νομίζω ότι είναι απόδειξη πολύ κοντής μνήμης εάν πει κανεί ότι πέρασε η κρίση και επομένως δεν ξανακοιτάμε πίσω και συνεχίζουμε με business as usual. Νομίζω ότι η καλύτερη κεφαλαιοποίηση της Βασιλείας και του Σέντερ 4 ε, βεβαίως δεν θα είναι η μοναδική απάντηση. Ε, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Στη διαχείριση κρίσης ε, θα μπουν και άλλα στοιχεία Γι' αυτό ε, ακριβώς εμείς έχουμε ξεκινήσει και άλλες ε, διαδικασίες ε, για τα παράγωγα, για τις ακάλυπτες πωλήσει. Παίρνουμε πάρα πολλές αποφάσεις και πάρα πολλά μέτρα. Κύριε Λαμπέρτσε, δύο λόγια για κάτι σημαντικό το οποίο αναφέρατε. Την τα μπόνους και τα μερίσματα. Αυτό το ζήτημα σαφώς ε, προβλέπεται ε, μέσω αυτού του ε, liquidity buffer και είναι σαφές ότι εάν η, τα ελάχιστα στοιχεία, οι ελάχιστες κεφαλιακές απαιτήσει δεν καλύπτονται, βεβαίως δεν θα έχουν δικαίωμα οι τράπεζες να δώσουν μερίσματα και μπόνους. Φυσικά, φυσικά ε, το κύριο μέλημά μα είναι να προστατεύσουμε τον κόσμο ε, και γι' αυτό θα ήθελα να σας καθησυχάσω κυρία Φόρντ ότι ε, πραγματικά αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Να, μην, να πληρώνουν οι τράπεζες για τι τράπεζε και όχι τελικά οι φορολογούμενοι πολίτες Επίσης, να σας πω ναι, στις διαπραγματεύσεις ε, της ε, ε, Βασιλείας καταφέραμε αυτό το ρυθμιστικό αποθεματικό ρευστότητας κατά 40% να αποτελείται από αυτές τις εγγυητικές επιστολές, τα lettre de έτσι ώστε να υπάρχει ε, πραγματικά μια, ε, να υπάρχουν αναθεωρημένα πρότυπα. Ε, όσον αφορά τώρα το business as usual, ξαναλέω ότι βεβαίως δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τις εξελίξεις στην αμερική γιατί το αμερικανικό σύστημα είναι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ ε, γιατί τα θέματα αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, εμείς παίρνουμε όλα τα μέτρα έτσι ώστε να μην πληρώνουν τελικά οι φορολογούμενοι αυτού του είδους της κρίσης. Κύριε Νίτρας, συμφωνώ, θέλουμε ενισχυμένη εποπτεία, γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο και μάλιστα και το Κοινοβούλιο τα μάλα έχει συμβάλει έτσι ώστε ε, να απαγορεύεται η χρήση τοξικών ε, προϊόντων. Τέλος, την κυρία ε, Ποδηματά να πω ότι για, τις, για αυτούς τους οργανισμούς της, της ικανότητας. Ναι, βεβαίως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτοί οι οργανισμοί. Θέλουμε ε, να αποφύγουμε αυτή την συγκέντρωση σε πολύ λίγα χέρια της δυνατότητας αξιολόγησης της αξιοληπτικής ικανότητας. Συζητήσαμε το θέμα αυτό και σε επίπεδο ε, Συμβουλίου Υπουργών και προωθούμε ε, τον, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα τροποποιήσει την υφιστάμενη κατάσταση. Τελειώνοντας να ξαναπώ ότι αυτά τα τρία στοιχεία επαναστάθμισης τα οποία αναφέρα προηγουμένως μας φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε κύριε Πίτρο Επίτροπε. Ε, κύριε έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως η συζήτηση ήταν σαφής, υπεύθυνη, με γνώσεις, νομίζω πως σχηματίστηκε μια καλή εικόνα. Και κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μετεχόντες και εσάς. Δεν αμφισβητούμε τη διαδικασία, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί θέσαμε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. ειδικά επί των πληγών εκείνων που προκάλεσαν οι τράπεζες με την κρίση ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία, απευθύνομαι συνάδελφο, αλλά η Βασιλεία προδικάζει το τι θα αποφασίσουμε. Οπότε γι' αυτό έπρεπε. Και βλέπετε, αν δεν κάναμε εμεί έκθεση ιδέα πρωτοβουλία, δεν θα υπήρχε καν συζήτηση. Οπότε πρέπει η Βασιλεία, η G20, όλου αυτού του νέου θεσμού που θα δημιουργήσουμε να είναι κοινοβουλευτικοί και δημοκρατικοί και να είμαστε ταυτόχρονα εμεί στην διαδικασία και όχι εκ των υστέρων να μαθαίνουμε τι γίνεται. Κυρίε και κύριοι, χρειαζόμαστε μια σχέση μεταξύ Βασιλείας 3 και διασφάλιστου Συστήματο. συστήματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν σύνδεση μεταξύ των δικών μας των αποφάσεων και της εφαρμογής παγκοσμίως, ειδικά στις ΗΠΑ. Θέλουμε να δούμε πριν ληφθεί η απόφαση ο, ποιος είναι ο ορισμός της ρευστότητα, ειδικά με βάση τους νέους νόμους της ΗΠΑ θα έχουν προβλήματα οι Αμερικανοί όσον αφορά τις εφαρμογές των νέων ε, προδιαγραφών ρευστότητος και προσπαθούν τώρα με νέα με νέες αξιολογήσεις, εξωτερικές αξιολογήσεις να εισαγάγουν εναλλακτικά κριτήρια. Είτε το ένα είτε το άλλο όμως, αλλά όχι και τα δύο για την Ευρώπη και μόνο ένα για τη ΣΥΠΑ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε, να επαγρυπνούμε και σας παρακαλώ κύριε Επίτροπε φροντίστε να κάνει τις μελέτες επιπτώσεων ή κομισιών και να τα πει αυτά και στους εθνικούς υπουργούς και στα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί η γνώση και η συνείδηση του τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα και τι σημασία έχουν αυτά στη Βασιλεία δεν υπάρχει στα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσουμε, να υπάρξει μια διαδικασία επικοινωνία και με τα εθνικά κοινοβουλία. Σα ευχαριστώ κύριε Καρά. Έληξε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριο Μπαρνία θα μείνει μαζί μα όλο το βράδυ. Τώρα είμαστε στη δήλωση τη Επιτροπή για την επιβολή προ